Ας αρχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Όσα ήθιστε, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Περνάμε στο πρώτο σημείο της μερίσιας διάταξης. Έγκριση της μερίσιας διάταξης. Σας έχει διανεμηθεί το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Προτείνω δύο τροποποιήσεις αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει και οι δύο γνωμοδοτήσεις που θα ψηφίσουμε σήμερα να πάνε στις αρμόδιες επιτροπές το συντομότερο δυνατό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις κατά τη διάρκεια της πρωινής μας συνεδρίασης, δηλαδή από τις 11 ως τις 12.30. Έχετε ενημερωθεί λοιπόν για την αλλαγή αυτή και μία ακόμα τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Βιαντόσκι μας ζήτησε να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή του για τις αιτήσεις εκθέσεις 2012-2013 για την αναλογικότητα και την επικορικότητα σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Να γίνει λοιπόν συζήτηση για τη γνωμοδότηση αυτή αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, δηλαδή αμέσως όταν ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Αν δεν έχετε λοιπόν αντιρρήσεις για τις δύο αυτές τροποποιήσει στη μέρη διάταξη, μπορούμε να εγκρίνουμε τη μέρη διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίρρηση. Σημείο 3 της σε διάταξη. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Σα ενημερώνω ότι ο εισηγητή για τη γνωμοδότηση για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών, νομισματικών και ρυθμιστικών ε, οργάνων. Είναι μια γνωμοδότηση που θα γίνει από τον Πάουλο Ρέιντζελ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να σας πω επίσης ότι σε σχέση με την ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου gender mainstreaming αρμόδια θα είναι η Constance Legrip από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξίσου να σας πω επίσης ότι μια ακρόαση για το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός αλλά και πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, μια ακρόαση που έχει να κάνει με την έκθεση Μπρέσο Μπρόκ και Φερχόφστατ, θα λάβει χώρα στις 26 Μαΐου από τις 9 ως τις 12.30 το πρωί. Ας περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις της Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών, Η συνεδρίαση των ιστών έγινε το πρωί. Τρία πράγματα έχω να σας πω. Πρώτον, συμφωνήσαμε ότι σε σχέση με την κατεξουσιοδότηση πράξη για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποφασίσαμε ότι Απριλίου 12 το μεσημέρι θα είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή συστάσεων ή ενστάσεων ή συστάσεων μη απόρριψης όσον αφορά την κατεξοδότηση αυτή πράξη σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού. Επομένως, οι συντονιστές σας θα σας ζητήσουν τη δική σας τη γνώμη και πρέπει να κινηθούμε αρκετά γρήγορα. Δεύτερον, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, τα δύο αυτά συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να υποβάλουν γνωμοδότηση για την έκθεση Mercedes Verhofstadt Brock Μπρέσο, με συγχωρείτε. Θα καλέσουμε λοιπόν τα δύο αυτά θεσμικά όργανα να υποβάλουν γνωμοδότηση και να συμμετέχουν ακόμα και στην ακρόαση που θα λάβει η χώρα στις 26 Μαΐου. Να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται διαπραγματεύσεις και εργασίες διαφόρων πολιτικών ομάδων για την ενδεχόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δύο συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την υψηλόβαθμη ομάδα, τον Αλάν Λαμασούγα και τον Κίφερ Χόφστατ. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλέσουμε τον Αλάν Λαμασούρ και τον Κίφερ Χόφστατ, τους συναδέλφους μας λοιπόν, σε μία συνεδρίαση προκειμένου να μας ενημερώσουν για τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτή την υψηλόβαθμη ομάδα εργασίας για την ανανέωση του, μάλλον την αναθεώρηση του συστήματο ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον βέβαια προκύψει επισήμω ένα τέτοιο σύστημα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όσον αφορά τη συνεδρία των συντονιστών. α περάσουμε τώρα στο σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που είχαμε στις 26 Φεβρουαρίου και στι 17 Μαρτίου. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά των δύο αυτών συνεδριάσεων και θεωρώ ότι εγκρίνονται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσια διάταξης. Θα καλύψουμε πολύ σύντομα το σημείο αυτό, καθότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την γνωμοδότηση που η δική μας Επιτροπή προετοιμάζει. Είχαμε συζήτηση και με τους συζητητές και με τους σκιώδες συζητητές και με διάφορους συμβούλους και καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λήψεις που καλύπτουν μέρος των τροπολογιών που έχετε καταθέσει. Υπάρχουν όμως και κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Νομίζω ότι έχετε και τον κατάλογο ψηφοφοριών. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη φάση αυτή, θα μπορέσουμε σε λίγο να προχωρήσουμε και με την ψήφιση της γνωμοδότησης αυτής. Να σας πω ότι ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ουσιαστικά υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων. Παρ' όλα αυτά εναπόκειται στους συντάκτες των τροπολογιών αυτών να μας πούνε αν θέλουν να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες που είναι κάπως εκτός δικής μας αρμοδιότητος. Γιατί ε, θα μπορούσαν ενδεχομένω να αφορούν την αρμοδιότητα άλλων ε, επιτροπών, των κανθήλων αρμόδιων επιτροπών. Σας δίνετε λοιπόν η δυνατότητα μέσω των τροπολογιών αυτών να εκφράσετε την άποψή σας Πάντως πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της δικής μας της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση να εναπόκειται σε εσά και στους δικούς σας τους συντονιστές να αποφασίσετε τι θα κάνουμε με αυτές τις τροπολογίες που είναι εκτός πεδίου εφαρμογή, εκτός αρμοδιότητος της δικής μας Επιτροπής. Ο κύριος Γκονζάλες Πώς θέλει να πει κάτι για τη δική του γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε λίγο αργότερα ή όχι. Νομίζω ότι έγινε μια επαρκή συνταλλαγή απόψεων, συζητήσαμε εκτενώς τη γνωμοδότησή σας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, Φάμπιο Μάσιμο Καστάλ, ο οποίο είναι ο συντάκτη γνωμοδότηση για την 30η και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε το έχετε το λόγο. Thank you very eh, Πρόεδρε, πολύ σύντομα, να σα παρουσιάσω πολύ σύντομα την γνωμοδότηση αυτή που έχει να κάνει με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, προσπάθησα να φερθώ στην σημαντικότερη προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουμε εμεί ω Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, αλλά και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ουσιαστικά να προωθεί την προβλεψιμότητα του κοινοτικού δικαίου και θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να γνωρίζουν με βεβαιότητα, διαφανή και γρήγορο τρόπο ποιε εθνικέ διατάξει, εφόσον υπάρχουν, θεσπίζονται κατά τη μεταφορά του ευρωνοσιακού δικαίου. Στη συνέχεια κάνω μια άμεση αναφορά στο διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο μέσω του οποίου θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται παρκώς για την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και πώς αυτή μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Στα πλαίσια της γνωμοδότησης αυτής, μολονότι αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις και έχει σημειωθεί πρόοδος μέσω τη θέσπισης του μηχανισμού EU Pilot, παρόλα αυτά εκφράζω και κάποιες ανησυχίες ή αναφέρομαι σε κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν, διότι η πλατφόρμα αυτή δεν είναι άμεσα προσβάσιμη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μάλλον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει ακριβώ ποιε είναι οι διαδικασίε επιπαραβάση τι οποίε επεξεργάζεται ή προτίθεται να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κατ' επέκταση και για τον Ευρωπαίο πολίτη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια άμεση πρόσβαση λοιπόν στο μηχανισμό αυτόν, να μην υπάρχουν άμεσες και έμεσες αρνητικές διαφορετικές μεταχειρήσεις. Επίσης, από την στιγμή που θεσπίστηκε η συνθήκη του Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί πλέον έναν σημαντικό συνομοθέτη, συμμετέχει πλήρως στα πλαίσια της ε, συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι συνομοθετεί για τα περισσότερα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό η ε, μεταφορά αυτή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία και η σχετική ενημέρωση για τη μεταφορά αυτή της κοινοτική νομοθεσία στην εθνική νομοθεσία να γίνεται με γρήγορο και άμεσο τρόπο και να μπορεί να ενημερώνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεώρησα λοιπόν ότι στους κόλπους των αρμόδων γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΥΠΟΛ, ΕΞΠΟΛ και Έρευνα, να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντικτύπου των βασικότερων ευρωπαϊκών διατάξεων που εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να παρακολουθούμε στο σύνολό του όλο τον νομοθετικό κύκλο. Κατά αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο αντίκτυπος της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και πώς μπορεί να βελτιωθεί κατ' επέκταση το νοσιακό δίκαιο. Θέλω να ελπίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα, μπορούς, θα μπορέσουν να συνταχθούν με την πρότασή μου αυτή και προφανώς είμαι διαλλακτικός για να ακούσω και τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων. Προσβλέπω λοιπόν να ακούσω τις δικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ Φαμπιό. Ο Τζότζο Σέπφλιν, ασκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καστάλτο για τη δουλειά που έκανα. Είναι πολύ διεξοδική κατά την άποψή μου. Έφεξε κάποια σημαντικά ζητήματα. Το θέμα της ασφαλείας δικαίου είναι ένα από αυτά. Πρέπει να είναι στο επίκεντρο των εργασιών μας. Γνωρίζαμε ότι με την πάρα του χρόνου βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει πάντα απόλυτη βεβαιότητα είναι κάτι που χρονικά είναι περιορισμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο τίθεται. Στη φάση που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να έχουμε στόχο τη μέγιστη δυνατή συνέπεια όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του κ. Καστάλντο, αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα της επιχρήσωσης του gold plating, δηλαδή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερφορτώνεται σε κάποια κράτη-μέλη και όχι σε άλλα κράτη, είναι κάτι που δημιουργεί ανώμαλες διαφορές, που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά είναι ανώμαλες οι διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Οπότε αυτό μειώνει την εμπιστοσύνη στα μάτια των πολιτών. Διότι κάνουν και συγκρίσει όχι μόνο τι γίνεται στη χώρα τους, τι γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη. Εγώ με κάποιους ε, Ούγγρους εκλογής είχα αυτή την εμπειρία. Το θέμα της διαφανείας επίσης είναι δύσκολο διότι ο νομικός κόσμος παράγει τη δική του ορολογία. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστεί σε κάτι που να είναι εύληπτο γενικότερα. Μπορούν να γίνουν βέβαια προσπάθειες, θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες. Και αυτό που σωστά έθεσε ο κύριος Κάσταλντο για το ρόλο του διαδικτύου είναι κάτι σημαντικό. Αλλά εκεί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Όταν μεταφράζεται η νομική ορολογία σε κάτι πιο εύληπτο ε, σε πιο ευρύτερο πλαίσιο αν διαστρεβλώνεται η γλώσσα αυτή. Ε, και κάποιοι ε, ειδικοί θα ξύνουν το κεφάλι τους στον αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, να διβάσουμε στον κόσμο ποια είναι η σημασία κάποιων νομικών πράξεων, νομικών πρωτοβουλίων Σημαντικό αυτό, από την άλλη όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν θα είναι ποτέ τέλειο, πάντα θα υπάρχουν κενά, Μπορώ να πω ναι στα άλλα που έθεξε ο κύριος Καστάλτο, ποια είναι η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν συνομοθέτου, η ανάγκη για πρόσβαση, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί τη λειτουργία του ε, και εξίσου σημαντικό είναι αυτό που αναφέρει όσον αφορά την εκ των υστέρων αξιολόγηση και τον ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά που έκανα. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές Ενρίκο Γκερέρο Σαλόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καστάλντο για το κείμενό του που μας παρουσιάζει και νομίζω ότι πετυχαίνει μια αρκετά σωστή ισορροπία όσον αφορά τις βελτιώσεις που επιφέρονται όσον αφορά το EU Pilot και που εντοπίζει τα κενά και την αδύναμη θέση στην οποία βρίσκεται το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το θέμα είναι πάρα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Καμιά φορά καθυστερώντας την ενσωμάτωση των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ε, υπάρχει μικρότερη περάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και υπάρχει μετά και υπερβολική ρύθμιση, το gold plating όπως αποκαλείται. Θα έπρεπε να μην ε, γίνεται ε, σκόπιμα εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών στα κράτη-μέλη. Έχουμε μια γνωμοδότηση. Ε, λοιπόν, είναι και το θέμα των, της διοργανικής συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών. Χρειάζεται μια διοργανική συμφωνία, λοιπόν, που θα έπρεπε να έχει τρία στάδια. Πρώτα απ' όλα την προετοιμασία, το νομοθετικό στάδιο και το στάδιο της αξιολόγησης. Θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση, να γίνει ένας προβληματισμός για να δούμε πώς εφαρμόστηκε η κοινοτική νομοθεσία, ποιος είναι ο αντίκτυπος για τους πολίτες και με ποιο τρόπο το θεσμικό μας όργανο, δηλαδή το Κοινοβούλιο, μπορεί να παρέμβει στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης. Το σύστημα EU Pilot μας επέτρεψε να παρέμβουμε στην αρχική φάση που δεν είναι φάση αξιολόγησης αλλά είναι η φάση καταγγελίας των παραβάσεων και έτσι δώσαμε μια φωνή στην κοινωνία των πολιτών και στο Κοινοβούλιο μέσω της υποβολής αναφορών στην Επιτροπή Αναφορών και μέσω άλλων εργαλείων να γίνονται καταγγελίες. Αυτό λειτουργήσε καλά, πρέπει να το πω αυτό. αποφύγαμε ε, πάρα πολλά προβλήματα αλλά δεν καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των παραβιάσεων. Αυτό που προτείνει ο κύριος Καστάλτο κατά την άποψή μου είναι κάτι συνεκτικό, δηλαδή το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, ε, το Κοινοβούλιο να μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι οι παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται το Κοινοβούλιο να έχει φωνή για την επίλυση των διαφορών, να είναι μια διέξοδος για επίλυση των διαφορών, αλλά αυτή είναι μια μικρή πετρούλα και μόνο. Και ευχαριστούμε τον κύριο Καστάλτο γι' αυτό. Αλλά η Επιτροπή μας, η Επιτροπή ΑΦΚΟ, θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη Διοργανική Συμφωνία, όπου όλες αυτές οι φτυχές και άλλες πτυχές πιστεύω θα παίξουν βασικό, σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος για την Άλτε. Για την Γκουε, ο Κώστας δεν είναι εδώ. Για τους πράσινους, Χωσέ Μαρία Τερικάμπρας, Μερσέντες Μπρεσό. Τα τακτικά μέλη, Μερσέντες έχει το λόγο. Ο Ρίτσαρτ. Α, είναι ο Ρίτσαρτ. Δεν θες εσύ Μερσέντες. Ο Ρίτσαρτ λοιπόν. Μετά, μετά εγώ. Εξαρτάται από αυτά τα απόλυτα, ο Ρίτσαρτ θα ήμουν συντομότατος, διότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκερέρο. Και πολλές από τις σοφές συστάσεις της εκθέσεως του κυρίου Καστάλντο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις της, για τη νέα διοργανική συμφωνία. Είναι μια ευκαιρία για μας για να προχωρήσουμε. Το άλλο σχόλιο που έχω είναι να επενέσω τον κύριο Καστάλντο. Σοφή προσέγγιση του, άκρος επικοδομητική που δεν το κάνουν πάντα τα μέλη της ομάδας τους στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ακολουθούν αυτήν την επικοδομητική προσέγγιση. Η εξαιρέσει επιβεβαιώνουν τον κανόνα, λέει η Πρόεδρος. Μεσέδες δεν θες να μιλήσεις. Γιατί να μην μιλήσω, λέει Μεσέντες. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καστάλτο για, την, ε, για το θετικό του αυτό έγγραφο. Πιστεύω και εγώ και πιθανότατα αυτό είναι ένα θέμα προς αντιμετώπιση στις εργασίες για, την, για το Better Legislation που για το Κοινοβούλιο θα είναι σημαντικότατο ζήτημα. Θα είναι σημαντικότατο να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που θα αφορά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική νομή Και υπογραμμίζω και στο επίπεδο των περιφερειών, διότι πολλές χώρες έχουν περιφέρειες που έχουν νομοθετική εξουσία. Όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, με την εξαίρεση της Γαλλίας πιστεύω, έχουν τέτοιες περιφέρειες με νομοθετική εξουσία. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ενσωμάτωση γίνεται σε τρία επίπεδα. Με τη δυνατότητα επιπλοκή τη καταστάσεω και να, τελικά να γίνεται αυτό το gold plating, η επιπλοκή τη νομοθεσία, με άλλα λόγια. Ε, σκεπτόμενοι τώρα ένα σημείο που αναφέρει στο έγγραφό του ο Ρίτσαρτ, το έγγραφο που ετοίμασε για την ομάδα μας, για το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Περιφερειακά Κοινοβούλια έχουν μεγάλο συμφέρον όχι μόνο να προωθήσουν τις πτυχές που αφορούν την επικουρικότητα, αλλά και τις άλλες πτυχές που αφορούν την ουσία της νομοθεσίας. Συνεπώς, για να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να δούμε και το ενδεχόμενο εκ των προτέρων συζητήσεις και επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων των καθήλων αρμοδίων επιτροπών για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Μία εργασία εκ των προτέρων που θα αφορά και τη μέθοδο αλλά κάποιες φορές και το περιεχόμενο. Αλλά το έργο όσον αφορά τη μέθοδο, πώς θα γίνεται αυτή η ενσωμάτωση είναι σημαντικότατο και ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Από τη δική μου εμπειρία έχω δει ότι όλα τα κοινοβούλια έχουν την τάση να περιπλέκουν την ομοθεσία είναι το παιχνίδι των τροπολογιών, των πολιτικών τοποθετήσεων και του του ρόλου. Και στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε νομοθεσία η οποία περιπλέκεται καθώς προωθείται και καμιά φορά ξεφεύγει και από τον βασικό επιδιωκόμενο στόχο. Λοιπόν, χρειάζεται εργασία για την απλούστευση, την νομοθετική, και πρώτα απ' όλα επαφών μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών φορέων. Εγώ θα υπογράμμιζα αυτό ότι σε πολλές χώρες, τις μεγάλες χώρες, νομοθέτες είναι δύο σε εθνικό επίπεδο. Εμείς πολύ συχνά το καλύπτουμε, το ξεχνάμε αυτό και μετά εκείνοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα διότι είναι πιο απόμακροι από τις επαφές που μπορούν να έχουν και συνομιλίες με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ Μερσέντες. Κύριε Σπλένκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ, Φάμπιο. Πολύ εμπεριστατωμένη η γνωμοδότησή σου για τις δύο εκθέσεις του 2012 και 2013 όσον αφορά την ετήσια παρακολούθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τρία σημεία θέλω να θίξω. και από τη σκοπιά ενό νέου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, και αυτά που θα πω νομίζω αφορούν όλου μα. Πρώτα απ' όλα, εμεί σαν Ευρωβουλευτέ, σαν ένα από του δύο συνομοθέτε, πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του εθνικού μα βουλευτέ στη διαδικασία εφαρμογή και Και γι' αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε μηχανισμούς, κοινούς μηχανισμούς και να μπορούν να υπάρχουν, να υπάρχουν κοινέ συνεδριάσει στι επιτροπέ ευρωπαϊκών υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων και να του εξηγούμε νομοθετήματα που εξετάζονται και κυρίω πώ αυτά, πώ οι οδηγίε ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο. Και μέχρι τώρα αυτή η προσπάθεια αυξάνει την ευαισθητοποίηση και κατανοούν καλύτερα ε, το νόημα που έχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό ευθυγραμμίζεται και με το πιλωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Ενώσεως για την καλύτερη νομοθεσία και του REFIT και προσπαθούμε να αποφύγουμε καθυστερήσεις στην εσωμάτωση εθνικό δίκαιο και να αποφύγουμε και ενδεχόμενες διαδικασίες κατά παράβαση. Και χαίρομαι ότι μέχρι τώρα είχαμε μόνο δύο υποθέσεις καθυστερημένης ενσωμάτωσης και το 2013 μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια διαδικασία κατά παράβαση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους σε αυτή τη μεταβατική φάση να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται, τόσο ώστε να υπάρχει και ευαισθητοποίηση και έγκαιρη, έγκαιρα να εφαρμόζεται ποιοτική νομοθεσία. Σχετικά με αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η γνωμοδότησή σου στέλνει τα σωστά μηνύματα, τα στέλνει και προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την υιοθέτηση των τελευταίων εκθέσεων που θα αφορούν τα δύο αυτά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που είπαν ότι η γνωμοδότηση που συζητούμε αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης. Τη συζήτηση για ένα νέο πλαίσιο διαθεσμική συμφωνίας. Οι προτάσεις, στάσει από τον εισηγητή και τον συγχαίρω για το έργο του αναφέρονται σε διαθεσμικές συμφωνίες και σε συζητήσεις σε σχέση με την νομοθεσία. Γίνονται κάποια πολύ γενικά σχόλια από τη μία πλευρά και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης της εφαρμογής των οδηγιών. Είναι το τελευταίο σημείο της γνωμοδότησης αυτό. Χρειαζόμαστε όμως ταυτόχρονα και διαθεσμική συνεργασία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη δικιά της αξιολόγηση, να αξιολογεί από μόνη της δηλαδή την εφαρμογή μιας οδηγίας. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να, κάνει, κάνουμε την ίδια δουλειά με την Κομισιόν. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης της εφαρμογής των οδηγιών. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Πράγκοβιτς. Συμφωνώ ότι πρέπει να γνωρίζουμε πώς εφαρμόζονται οι οδηγίες. Ναι, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες. Πώς μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να επηρεάσει τη διεργασία εφαρμογής. Γιατί έχω αυτές τις αμφιβολίες. Τα περισσότερα νομοθετήματα τα οποία εφαρμόζονται μέσω οδηγιών ε, είναι ουσιαστικά ε, πρωτοβουλίες των εθνικών κοινοβουλίων. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τρόπον την ένα δευτερεύοντα ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Έρχονται δηλαδή μετά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Άρα, πώς μπορούμε να ενεργήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να έχουμε γνώσεις και σύστημα αξιολόγησης ώστε να ξέρουμε πώς εφαρμοζόνται αυτές οι οδηγίες και χρειαζόμαστε και ένα σύστημα αξιολόγησης των καθυστερήσεων συχνά υπάρχουν ε, σημαντικά θέματα. Παραδείγματο χάρη οδηγία για το λαθρεμπόριο των ανθρώπων δεν έχει εφαρμοστεί από πολλέ χώρε. Ο επόμενο ομιλητή. Ε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κασαλτό, αλλά έχω κάποια ερωτήματα σε σχέση με την παραγράφο 2 και 4. Λέτε στην παραγράφο 2 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις. Τι θέλετε ακριβώς να πείτε. Και στο 4 ζητάτε ένα σύστημα για την αξιολόγηση ex post των, αντικτύπων. Και σύμφωνα με τη νο, σύνηθη ε, νομοθετική διαδικασία. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν θα είναι χρήσιμο αυτό το ε, μέσο το οποίο προτείνεται. Υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν να το ζητά. Φάβιο, σου ξαναδίνω το λόγο. Α, η Κομισιόν, η Κομισιόν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον το οποίο ε, δείχνεται για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου ε, πολύ σημαντικά ζητήματα έχουν τεθεί. Πώς εσύ, σαν, εσείς σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή μπορείτε να συμμετάσχετε στην προώθηση αυτού του σημαντικού ζητήματος στα κράτη-μέλη. Βεβαίως θα μιλήσουμε για τη διαθεσμική συμφωνία, είναι ένα ζήτημα προς διαπραγμάτευση αργότερα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται απόλυτα να συνεργαστεί μαζί σας και να εξετάσει τις δυνατότητες της αποτελεσματικής εφαρμογής εκ μέρους όλων των θεσμών που εμπλέκονται. Και βεβαίως η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Τούτου λεχθέντος δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια τώρα σε σχέση με τα διάφορα σημεία, τα οποία βεβαίω θα εξετάσουμε με προσοχή και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Φάμπιο, έχεις το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο και είπαν ότι είναι καλή εργασία που έχω κάνει. Όλους αυτούς οι οποίοι λοιπόν εκτιμούν την εργασία μου. Λαμβάνω βέβαια υπόψη και όλες τις παρατηρήσεις ξεκινώντας με τον κύριο Σέμπλιν. Νομίζω ότι και αυτός αλλά και ο κύριος Γκερέρο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ επικοδομητικές παρατηρήσεις. Ως Ιταλός γνωρίζω ότι στη δική μου τη χώρα υπάρχουν πολλές διαδικασίες ή παραβάσεις που είναι ακόμα ανοιχτές. Και όπως είπατε και εσείς αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων πρέπει να συμβάλλουμε πολύ στο να θεραπεύσουμε την κατάσταση. Επίση, η νομική ασφάλεια είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ είμαι νομομαθή, συμφωνώ μαζί σα. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας διτός διάβλος επικοινωνίας. Να υπάρχουν δηλαδή κάποιες υποχρεωτικές πληροφορίες στις οποίες να έχουμε πρόσβαση και οι οποίες μπορούν να είναι και τεχνικές, αλλά από την άλλη να μπορούμε να έχουμε και μια κάποια γλώσσα λίγο πιο εκλαϊκευμένη, προκειμένου ο μέσω Ευρωπαίου πολίτη να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν και έναν διάβλο επικοινωνίας και ενημέρωση, ο οποίο θα είναι λίγο πιο απλουστευμένο και θα έχει και ένα χαρακτήρα κάπω παιδαγωγικό και εν τέλει θα φέρνει πιο κοντά τον Ευρωπαίο πολίτη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσον αφορά τα όσα είπε ο συνάδελφος Γκερέρο, συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα μικρό βήμα. Νομίζω θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας, θα πρέπει να διευρύνουμε τη σκοπιά μας. Προφανώς δεν μπορούμε εμείς να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο όλο σύστημα μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την κεντρική σημασία που πρέπει να έχει μια διοργανική συμφωνία. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο στέλνουμε και το οποίο πρέπει να στείλουμε και μας έχει απασχολήσει αυτό και σε προηγούμενες ε, συνεδριάσεις ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να πάει προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να εμβανθύνουμε την όλη συζήτηση για το ρόλο που πρέπει να έχουμε εμεί ω θεσμικό όργανο, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα από του Ευρωπαίου πολίτε. Επομένω, βρισκόμαστε εμεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, πολύ πιο κοντά στον ίδιο τον Ευρωπαίο πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βοηθάμε και εμεί τη βελτίωση τη προσβασιμότητα προς τις πληροφορίες αυτές. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Κόρμπετ, καθώς επίσης και τη συνάδελφο Μπρέσο για τα θετικά του σχόλια. Η κυρία Μπρέσο πριν από λίγο αναφέρθηκε στα περιφερειακά τοπικά κοινοβούλια και ότι όντως υπάρχει μια πολυεπίπεδη κοινοβουλευτική διαδικασία σε διάφορα κράτη-μέλη. Και όντω ε, έχετε δίκιο, στη Γαλλία ακόμα έχουμε ένα πολύ πιο κεντρικό σύστημα. Δεν υπάρχει αυτή η διαβίβαση κοινοβουλευτική αρμοδιότητα σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο όμω κάτι τέτοιο ισχύει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη μα και να βρούμε κάποιε κατά περίπτωση λύσει προκειμένου να μπορούν και τα τοπικά κοινοβούλια, οι εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Και νομίζω ότι σε αυτό αναφέρθηκε και ο συνάδελφο Πλάνκοβιτ Να μπορέσουμε δηλαδή να θεσπίσουμε έναν τρόπο, αν μη τι άλλο άτυπο, ανεπίσημο, προκειμένου να μπορούν να ενημερώνονται καταλήλως και τα περιφερειακά κοινοβούλια, τα τοπικά κοινοβούλια και να μπορούν να συμμετέχουν έστω και άτυπα, έστω και ανεπίσημα την όλη διαδικασία νομοθετική που διεξάγεται εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συμβάλλουν και τα τοπικά κοινοβούλια στην πιο άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά του κοινοτικού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Ξέρω ότι για παράδειγμα υπάρχει μια επιτροπή της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά και ουσιαστικά είχαμε συζητήσει όταν συμμετείχα εγώ στην επιτροπή αυτή την ε, δυνατότητα αυτή να μπορούμε να επεμβαίνουμε ως Επιτροπή Εθνικού Κοινοβουλίου σε συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε φορά που συζητούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, μεταφορά του ενωσιακού δικαίου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προτείνουμε ένα κάποιο μοντέλο, θα μπορούσαμε να βασιστούμε ενδεχομένω και σε αυτό το ιταλικό παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει και για άλλα κράτη-μέλη. Ο συνάδελφος Ζιαντόσκι, ελπίζω ότι προφέρω σωστά το όνομά σας, αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όντως θα πρέπει να υπάρχει μια διοργανική συνεργασία και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δυστυχώς όμως, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η συνεργασία αυτή διοργανική δεν ήταν πάντα τέλεια και αποτελεσματική. Διαφορετικά δεν θα βλέπαμε και στη γνωμοδότησή μου όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία εκφράζουμε σε σχέση με την κατάλληλη και πιο έγκαιρη πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς υστερεί ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις δυνατότητες που του δίνονται να ενημερώνεται. Πάντως, πρέπει στα πλαίσια της συζήτησης που θα γίνει για τη Διοργανική Συμφωνία να θίξουμε και το ζήτημα αυτό από τη δική μου την πλευρά δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα και η δική μου η πρόταση δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαστικά πανάκια και ότι θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς προτείνω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αυτόν τον αυτόνομο ανεξάρτητο μηχανισμό. Πάντως ε, προσβλέπω και στις δικές σας περαιτέρω παρατηρήσεις και να δούμε τι έχουν να πούνε και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τα οποία ασχολούνται με το ζήτημα της μεταφοράς του νοσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Πάντως θα μπορούσαν να γίνουν και από εσά πιστεύω και κάποιες άλλες προτάσεις προκειμένου να καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια καλύτερη πρόταση, πιο πλήρη από αυτή την οποία προτείνω εγώ. Νομίζω ότι η δυνατότητα αυτή θα μας δοθεί και στην συζήτηση που θα γίνει με τους κοιόδης εισηγητές. Πάντως είμαι απόλυτα διαλλακτικός και ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση ενδεχομένως να προτείνεται. Και να ολοκληρώσω δίνοντας αυτές τις δύο διευκρινήσεις ε, που ζήτησε ο συνάδελφος Τζο Λάιν Νομίζω ότι ε, ήδη απάντησα για το σημείο 4 της γνωμοδότησης. Αναφέρθηκα δηλαδή μόλις τώρα σε αυτή την πρόταση ανεξάρτου συστήματος εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά το ζήτημα της άμεσης ή έμεσης διάκρισης που αναφέρω στη γνωμοδότησή μου. Θεωρώ ότι όντως υφίσταται διακριτική μεταχείριση διότι όταν γίνεται ο διάλογος στα πλαίσια του EU Pilot ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαίο πολίτη, πολύ συχνά ο Ευρωπαίο πολίτη καταλήγει να μην γνωρίζει τελικά αν μια συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί ή όχι στην εθνική νομοθεσία ή αν έχει μεταφερθεί ελλιπώς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε για τον Ευρωπαίο πολίτη μια καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και θα μπορούσε αυτό να γίνει και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο το οποίο αποτελεί έκφραση, αν θέλετε, της λαϊκής βούλησης. Είναι άμεσα εκλεγμένο από τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα μπορούσε λοιπόν να συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μειωθεί αυτό το έλλειμμα πληροφόρησης, το έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει πολλές φορές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ επικοδομητική αυτή συζήτηση που είχαμε και καταφέραμε πολλές φορές στα πλαίσια της συζήτησης αυτής να καλύψουμε και πολλά περισσότερα θέματα από αυτά που προβλεπόταν στα πλαίσια της γνωμοδότησης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Είμαστε χαλαροί όσον αφορά τις προθεσμίες για τροπολογίες. 4 Μαΐου μπορούμε να το ορίσουμε, αν θέλετε. 5 το απόγευμα, 6 το απόγευμα, 5 το απόγευμα. 1η Μαΐου. Νομίζω 4 Μαΐου είπε και τελικά η κυρία Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ επικαδομητική. Και τώρα ε, περνάμε στο, στην ψηφοφορία, όμως πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 11. Έχουμε 8 λεπτά ακόμη μέχρι τις 11. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε όμως την ψηφοφορία πριν από τις 11. Dear colleagues, I think we have to start the, the, vote. Πρέπει να ξεκινήσουμε ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε δύο θέματα. Το TTIP πρώτα και μετά το έψι. Θα ελέγξουμε πρώτα όμως πώς λειτουργούν τα μηχανήματα και οι κάρτα σας. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία να δούμε πώς λειτουργούν τα μηχανήματα, αν λειτουργούν σωστά. Somebody Υπάρχει κάποιος χωρίς κάρτα. Έγινε ψηφοφορία στην νομική επιτροπή, ξέχασα την κάρτα μου, αλλά θα έρθει ένα λεπτό περίπου. Θα σας περιμένουμε, λέει η Πρόεδρος. Έρχεται, έρχεται, καταφέρνει. You don't have. No, you, do. Έχετε, δεν έχετε. Α, απλώς υποστηρίζετε τον συνάδελφό σας. Εντάξει.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 Does all these decisions, it says that chair, committee, if there is another objection. Yes. es una enmienda de compromiso sí. no aceptada por el reportero. Sí, sí. Uh, so I, I think everybody's here and everybody's is. Uh... Ήρθατε όλοι. Είστε έτοιμοι. Μα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έχουμε την ψηφοφορία για το TTIP. Ξεκινάμε τροπολογία 1 υπέρ. Τροπολογία 1 υπέρ. Uh, sorry. Α, υπάρχει ακόμα πρόβλημα.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 Συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν το γνώρισα. Υπήρξε κάποιο αίτημα του εισηγητού για το TTIP να ψηφίσουμε δεύτερο το θέμα του TTIP. Εντάξει, δεν κάνει διαφορά. Όσον αφορά την μερίσια διάταξή μας, ζητώ συγγνώμη. Οπότε πάμε αμέσως στην άλλη ψηφοφορία για το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Στρατηγικών Επενδύσεων. Ακολουθούμε διαφορετική σειρά. Για τεχνικούς λόγους. Αλλάζουμε. Δεν το γνώριζα. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το ΕΦΣΙ. Πρώτα. Πρώτα το ΕΦΣΙ. Ψηφίζουμε το ΕΦΣΙ. Τροπολογία 86 υπέρ κατά, αποχές. Έλμαρ, έχεις αίτημα που είναι αντίθετο από το αίτημα της ομάδας σου, κουβέντιας, έπαν το έχεις κουβεντιάσει με το συντονιστή σου πριν. Προχωρούμε, προσπαθούμε πάμε γρήγορα. Τροπολογία 86 την ψηφίσαμε, εγκρίθηκε. Τροπολογία... Βλέπετε σε τι ομάδα είμαι, απίστευτο. 87 υπέρ. Τροπολογία 87 υπέρ. Who, who is in favor? He will come, he will come. Okay, don't. No, we have one. Amendment 87. Τροπολογία 87. Ποιος είναι υπέρ? Είναι κάποιος που είναι υπέρ της 87? No. Who's against? κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 89 υπέρ κατά έλεγχος για την 89 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία για την 89 The Πέρας σου. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 89 εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 90. 90. 9. 90. Πέρας. Το ΕΛΚ έχει μια ψήφο παραπάνω. Μόνο ένα άτομο να βγάλει την κάρτα του, γιατί πολλές φορές βγάζουν όλη την κάρτα τους. Ας βγάλει ένα άτομο την κάρτα του παρακαλώ το ΕΛΚ. Τζόρτζ, σε παρακαλώ να αποσύρεις την κάρτα σου. Έτσι για ένα δευτερόλεπτο σου παρακαλώ. Βγάλ την κάρτα σου. Ο κύριος Πλένκοβιτς έβγαλε την κάρτα του. Ο Τζόρτζ ξαναβάζει την κάρτα του σου. Ωραία, καλά είμαστε τώρα. Ψηφίζουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία, απερίφθη μάλλον. 15-9 απερίφθη. Uh, any problem? No, it was rejected already. Απερίφθη, απερίφθη. 91, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και για την 91, άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει κάποιος, δεν πειράζει, πέρας, απορρίπτεται. 92 υπέρ 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υπολείπτεται σαφώς 13 υπέρ κατά έλεγχος γιατί 13 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ενενήντα πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα 96. Να σας ενημερώσω για κάτι. Σχετίζεται με τη 41, την 99, 102 και 103. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί λοιπόν. Αν εγκριθεί όλες εγκρίνονται, αν απορριφθεί αυτή απορρίπτονται και οι υπόλοιπε, οι συναφεί. Ψηφίζουμε την 96 που αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα τροπολογιών υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται Εκατόν τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 αποσύρεται 110 υπέρ 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κατά τμήματα για την 118 πρώτο τμήμα της 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασ... απορρίπτεται απερίφθη 119 συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 απεσύρθη συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται ας γίνει έλεγχος για την 129 Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 Μόνο ένα τμήμα έχουμε στην 136, το άλλο τμήμα καλύπτεται από τη συμβιβαστική. Ε, με την επιφύλαξη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τι, ξέχασα κάτι. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν 139 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 140 υπέρ α έχει αποσυρθεί μάλιστα μάλιστα 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σαφώς 142 υπέρ κατά έλεγχος για την 142 Πέρας. Απορρίπτεται. 143. Απεσύρθη. 144. 144 υπέρ. Κατά. Μικρή διαφορά. Έλεγχος για την 144. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Δεν ξεκίνησα. Mm. Κάποιος μας παρακολουθεί εδώ πέρα. Λοιπόν, ακόμα κάποιοι ψηφίζουν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 148 απεσύρθη, 149 ψηφίζουμε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Δεν είναι μόνο αρμοδιότητες ΣΑΦΚΟ και είχαν οι συνάδελφοι δικαίωμα να αφήσουν τις τροπολογίες και να τι αποσύρουν αν θέλουν να ψηφιστούν. 150 λοιπόν υπέρ κατά Ήταν σαφές το αποτέλεσμα 150 λέει πρόεδρος. Μπορούμε να ελέγξουμε αν θέλετε, αν έχετε αφιβολίες. 150 ηλεκτρονικός έλεγχος. 150. πέρα ψηφοφορίας. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, δίκιο είχατε. Πρέπει να επαγρυπνούμε. 151 καταπίπτει. 152. Ψηφίζουμε το 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Μπορούμε να κάνουμε μέχρι 164 όλες μαζί. Συμφωνείτε. 155 και 164 μαζί. Όλες μαζί. 155, 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 καταπίπτει. 100 66 ψηφίζουμε υπέρ κατά κατά παρακαλώ εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ας γίνει ένας έλεγχος για την 167 It was 167. We close the vote. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170, 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Την 170 επαναλαμβάνω. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελήξη απορρίπτεται 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ. Κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 171. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 12 προς 11. 172. 173, καταπίπτει 172. 174 μάλλον, υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Ηλεκτρονικά λοιπόν την 174. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. 176 υπέρ. Κατά. Ε, ελέγχουμε το 176. Ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177-178. Καταπίπτουν όχι το 178 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές 181 υπέρ κατά ελέγχουμε την 181 Έληξη ψηφοφορία απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ Έλμαρ 28 Το πρόβλημα είναι να ξεχάσουμε να ψηφίσουμε κάτι 28 υπέρ Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. 28 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Για την 28. Έλξη ψηφοφορία εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική έξι. υπέρ. Α, την 185 δεν ψηφίσαμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική έξι. υπέρ. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά δεν ξέρω. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Έληξη ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Ε, τέτοιο μείγμα. 190 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ούτε οι ομάδες το ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο σήμερα. 190 ηλεκτρονικά έληξε η ψηφοφορία ένα, ε, ένας ΕΛΚ παραπάνω εντάξει τώρα ωραία γκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές Εκ... απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 είναι το επόμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά και τα λοιπά εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το επόμενο αποσύρεται, πάμε στο 203, υπέρ. Διακόπτη πρόεδρος. 203 με 207 μπορούμε να ψηφίσουμε όλα μαζί. Ωραία. 203 με 7 οι σοσιαλιστές λένε ναι. Υπέρ. Κατά αποχές 208 ε, με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά απορρίπτεται 212 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για το T212. Πλησιάζουμε στο τέλος, μην ανησυχείτε. Έληξη ψηφοφορία, απορρίπτεται το 212. Το 213 το ψηφίζουμε τώρα, υπέρ, κατά. Δεν ξέρω. ηλεκτρονικό έλεγχος, λέει η πρόεδρο. Έληξε. Απορρίψετε. Τώρα ερχόμαστε στα citations. Ένα. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Ένα. Υπέρ εγκρίνεται 34 υπέρ κατά ...35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά δεν ξέρω ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ λίγη ψηφοφορία ένα ΕΛΚ πρέπει να αποχωρήσει από την ψηφοφορία απορρίπτεται 40 υπέρ κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά δεν ξέρω ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ οι σοσιαλιστές να ψηφίσουν παρακαλώ μαζί με τους έλκος και έτσι θα διευκολυνθούν τα πράγματα δεν θα έχουμε κλιμακώσεις κλείνουμε την ψηφοφορία Απορρίπτεται. 43 υπέρ. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για το 48. Έλλειψη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 αποσύρεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ να ελέγξουμε την 52 σας παρακαλώ ηλεκτρονικά λήξη πέρας Απορρίπτεται. 53 υπέρ. 53 υπέρ κατά. η κατάσταση. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δύο ΕΛΚ παραπάνω από τον λογικό αριθμό. <laughs> Απεσύρθησαν. Ωραία. Ε, ποτέ δεν τελειώνουμε με τους ΕΛΚ. Έχουμε πλεόνασμα. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Δύσκολοι συνασπισμοί να ποσοτοτικοποιηθούν. Δύο ψηφίζουν παραπάνω. Εντάξει είμαστε τώρα. Απορρίπτεται 56 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε όμως καλύτερα. 56. Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Νομίζω την ίδια κατάσταση. Θα ψηφίσουμε και το 57 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 57. Ένα ΕΛΚ παραπάνω από τον κανονικό αριθμό. Έλξη ψηφοφορία. απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61. Έλεξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 4. Έλμαρ 4. Υπέρ. Κατά. Ο Έλμαρ πρέπει να ε, κάτσει μόνος του σε μια γωνία τιμωρία. Είναι απίθανο. Κρίθηκε τώρα τι έγινε. Ποιος είναι υπέρ της 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Α, καταπίπτει, καταπίπτει 62. Παίρναμε στην 63. Κατευθείαν. Ψηφίζουμε την 63 σας παρακαλώ, υπέρ κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Παρακαλώ για την 63. Άντε, πλησιάζουμε. <laughs> Απορρίπτεται. 64 καταπίπτει. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά Ελέγχουμε την 65 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Έλξη ψηφοφορία. Ένα ΣΕΛΚ παραπάνω. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά δύσκολο ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 68 παρακαλώ έλξη ψηφοφορία εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά τι κάνανε οι σοσιαλιστές δεν πρόσεξα λοιπόν την 70 παρακαλώ την ελέγχουμε έλεξη ψηφοφορία ηλεκτρονικά 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 εφαναρχόμαστε στην 71 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ Έληξη ψηφοφορία Απορρίπτεται, Έλμαρ, έχεις δίκιο. Το ένστικτό σου είναι σωστό. 73, υπέρ. Κατά, αποχές. Γκρίνεται. 72, καταπίπτει. 74, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 75 75 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται, όχι, όχι. Ε, καμιά φορά σηκώνετε το χέρι σας πολύ γρήγορα, τα κατά μαζί με τα υπέρ και μπερδεύομαι. Ας το ελέγξουμε καλύτερα, λέει η Πρόεδρος. Την τροπολογία 75 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. 10 υπέρ εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά από ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 81 Έληξη ψωφού ψηφοφορία απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 83 υπέρ. έχουμε ηλεκτρονικά. Την 83. Πέρας. Απορρίπτεται 84 υπέρ. 10 προς 14 περίπου. 84 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 84. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 προς 12. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα ΣΕΛΚ παραπάνω. Ένας να αποσύρθει παρακαλώ, ένας. Ε, εντάξει είμαστε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 8-3-3. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 18 υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ας έχετε μπροστά σας τον κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα για το TTIP. Έλμα, είσαι και εσύ έτοιμος. Γι' αυτό δεν ήρθες, για το TTIP. Εκτός μικροφώνου, κύριος Μπρόκ. Καθυστέρησες, αλλά έχεις τους λόγους σου. Λοιπόν, τροπολογία είναι υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας ανακατά. Ήχος. Έχουμε πάλι μία επιπλέον ψήφα από το ΕΛΚΑ. Διευθετήθηκε όμως εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά μάλλον άρθρη ψηφοφορία για την τροπολογία 4 πέρας εγκρίνεται 12 υπέρ 11 κατά τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 15. Υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 2. Εδώ πέρα έχει προκύψει το εξή ζήτημα. Έχουμε την προτινόμενη αυτή από τον εισηγητή συμβαστική τροπολογία παριθμών 2, η οποία καλύπτει διάφορες τροπολογίες Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Χθε όμως, χθε το απόγευμα, έγινε μία άλλη πρόταση συμβαστικής τροπολογίας, σύμφωνα με την οποία, δεν ξέρω καν ποιος την κατέθεσε, οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές και οι γκουε, όχι οι πράσινοι και οι γκουε κατέθεσαν αυτή την άλλη συμβαστική τροπολογία, Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 174 του κανονισμού μπορούμε να ψηφίσουμε και αυτή την επιπρόσθετη συμβαστική τροπολογία, μολονότι υποβλήθηκε μετά την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, ξέρετε ότι μπορούμε να καταθέτουμε συμβαστικές τροπολογίες και αργότερα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία, την αρχική του εισηγητή και στη συνέχεια, αν εγκριθεί αυτή η συμβαστική τροπολογία, η πρώτη ή άλλη καταπίπτει, και θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και τις επιπρόσθετες τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τη συμβαστική τροπολογία 2. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Υπάρχει αντίρρηση. Ε, μια ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Τι θα γίνει αν καταπέσουν και οι δύο συμβαστικέ τροπολογίε. Θα ψηφίσουμε όλε τι υπόλοιπε τροπολογίε. Ναι. Αν οι δύο συμβαστικέ τροπολογίε καταπέσουν, θα ψηφίσουμε τι υπόλοιπε τροπολογίε. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία της πρώτης συμβαστικής τροπολογίας 2 του εισηγητή. Διακόπτη πρόεδρος. Ο κύριος Ντιόν έχει το λόγο. Δεν γίνεται να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες, τις επιμέρους τροπολογίες πριν τις συμβαστικές. Την τροπολογία 16 τουλάχιστον. Γιατί άλλωστε η τροπολογία 16 είναι μια τροπολογία που ζητά την απόρριψη της πρότασης. Επομένω, αν απορριφθεί η πρόταση αυτή, δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε την υπόλοιπη συζήτηση και ψηφοφορία. Μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή την τροπολογία 16 που ζητά την απόρριψη του κειμένου, τη διαγραφή του κειμένου. Πρόεδρο. κοιτάξτε, αποφασίσαμε, αποφασίζω μάλλον ω πρόεδρο, ότι θα ψηφίσουμε πρώτα τι συμβαστικέ τροπολογίε και μετά τι επιμέρου τροπολογίες. Έτσι προχωράμε συνήθω.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 Ο εισηγητής ε, έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία, κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για ένα ολόκληρο μήνα, μίλησε με όλους τους σκιώδεις εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες μέχρι χθε το βράδυ. Καταφέραμε λοιπόν να διασφαλίσουμε μια πλειοψηφία που καλύπτει τις περισσότερες πολιτικές ομάδες και καταλήξαμε σε αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Τώρα βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή υποβλήθηκε μια άλλη συμβαστική τροπολογία χωρίς να έχει ενημερωθεί καν ο Νομίζω ότι δεν μιλάμε για ορθή κοινοβουλευτική πρακτική. Είναι αθέμητο να γίνεται κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι είναι αθέμητο κατά αυτόν τον τρόπο να προσπαθείτε να παραγωνίσετε τον εισηγητή ή να παρακάμψετε τη δική του τη συμβαστική τροπολογία. Εργάστηκε πολύ σκληρά για ένα ολόκληρο μήνα ο εισηγητής, πρόεδρος. Μα γι' αυτό σας είπα ότι πρώτα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία και θα δούμε τι θα κάνουμε με την επόμενη. Λοιπόν, ξεκινέψω φορέα για τη συμβαστική τροπολογία 2, την αρχική του εισηγητή. Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ονομαστική ψηφοφορία, όχι ηλεκτρονικά, ονομαστική ψηφοφορία. Uh, we, don't have yet everybody, so we keep vote open. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε ότι όλοι συμμετέχουν. Αναφερόμαστε, ψηφίζουμε την αρχική συμβαστική τροπολογία παριθμών 2 του εισηγητή πέρας της ψηφοφορίας, προτού βάλει κανείς άλλο στην κάρτα του, και απορρίπτεται. Can we the, But did they, did they ask? Yeah, okay. So now, the, the, now we go to vote the other. Περνάμε στην ψηφοφορία της επόμενης συμβαστικής τροπολογίας. Πρέπει να ξεκινήσει η ψηφοφορία και για τη δεύτερη αυτή συμβαστική τροπολογία. Λοιπόν, Άρτη ψηφοφορία για τη δεύτερη συμβαστική τροπολογία. Ψηφίζουμε τώρα την δεύτερη συμβαστική τροπολογία. Ωραία, πέρας. Εγκρίνεται. 12 υπέρ 11 κατά. Συνεπώς δεν θα ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες, διότι η δεύτερη συμβαστική τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες αυτές που θα ψηφίζαμε. Περνάμε στη τροπολογία 28. Ή λυπάμαι, όλε οι υπόλοιπε τροπολογίε καταπίπτουν γιατί καλύπτονται από την δεύτερη συμβαστική τροπολογία που μόλι ψηφίσαμε και εγκρίναμε. Δεν είναι συμβατή τροπολογία που ζητάτε. Compatible. Yeah. No, but the, the problem with 16 is that it is not... Δείτε, η τροπολογία 16 δεν συνάδει με τη συμβαστική τροπολογία 2 που μόλις ψηφίσαμε. Δεν είναι συμβατή. Δεν καλύπτεται μεν, αλλά δεν είναι και συμβατή, άρα καταπίπτει. To inclusion. Yeah, yeah, but I'm saying this.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 Είμαι απόλυτα εξοικειωμένο με αυτά τα οποία ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί με έχουν απασχολήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κείμενο το οποίο εγκρίναμε δεν συνάδει, δεν συνάδει με τις τροπολογίες τις οποίες ψηφίσαμε. Ο, η τροπολογία που καλούμε θα αυτή τη στιγμή να ψηφίσουμε, που ζητάει ο κύριος Ντιογόν, ουσιαστικά διαγράφει, ακυρώνει το μέσο αυτό το οποίο θέλουμε να εγκρίνουμε και το οποίο μόλις εγκρίναμε μέσω της συμβαστικής τροπολογίας. Αναφέρομαι στο Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους, ISDS. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Επίσης, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα. Δεν γίνεται να ψηφίζουμε μια συμβαστική τροπολογία και εκ των υστέρων να λέμε ότι υπάρχει μια άλλη τροπολογία η οποία δεν καλύπτεται ή δεν είναι συμβατή. Νομίζω ότι αν θέλετε να ψηφίσουμε μια τροπολογία ξεχωριστά, θα πρέπει αυτό να λέγεται εκ των προτέρων. Δεν γίνεται να κάνουμε μια, συμβαστη... μια ψήφιση, μια ψηφοφορία για συμβαστική τροπολογία και εκ των υστέρων να λέμε ότι υπήρχε τροπολογία η οποία δεν καλυπτόταν από τη συμβαστική τροπολογία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιο προηγούμενο. Όχι, λέει ο Πρόεδρο, για μένα η τροπολογία 16 ουδέποτε καλυπτόταν από τη συμβαστική τροπολογία. Πηγαίνει στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Ουσιαστικά η συμβαστική τροπολογία θέλει να δημιουργήσει ένα μόνιμο μηχανισμό επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου. Αναφερόμαστε εδώ πέρα ίσως στην μακροπρόθεσμη λύση δημιουργίας ενός διαιτητικού δικαστηρίου, ενώ η τροπολογία 16 προτείνει τη χρησιμοποίηση των εθνικών δικαστηρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δύο τροπολογίες δεν συνάδουν, δεν είναι συμβατές, είναι για μένα σαφές αυτό. Ποιος, ε, ποιος πρέπει να πάρει τώρα πρώτο το λόγο, κυρία Περβόνς Μπερές. Να εξηγήσω ενδεχομένω την κατάσταση, να μου δώσετε λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αν υφίσταται αυτή τη στιγμή κάποια αμφιβολία όσον αφορά το ζήτημα αυτό, μήπως θα έπρεπε δημοκρατικά να ψηφίσουμε. Αν υφίστανται λοιπόν αμφιβολίες όσον αφορά το ζήτημα αυτό και συγκεκριμένη τροπολογία, δεν θα έπρεπε μάλλον να την ψηφίσουμε. Αυτή είναι η πιο δημοκρατική επίλυση του ζητήματος, κυρία Πρόεδρε. Ας ψηφίσουμε την τροπολογία 16. Και αν απορριφθεί, απορρίφθηκε. Αν εγκριθεί, εγκρίθηκε. Κυρία Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Είμαι συντάκτης της ε, τροπολογίας αυτής. Να σας πω πώς έχει κατάσταση. Στον κατάλογο ψηφοριών επίσης βλέπω ότι αν είχαμε ψηφίσει τη συμβαστική τροπολογία 2 την πρώτη εκδοχή του συντάκτη γνωμοδότησης, τότε εκεί λέγεται ξεκάθαρα ότι αυτή η συμβαστική τροπολογία δεν καλύπτει τις τροπολογίες 16, 17 και κάποιες άλλες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια παρόμοια κατάσταση γιατί η δεύτερη εκδοχή της συμβαστικής τροπολογίας ουσιαστικά ξεκινάει, ανοίγει το ίδιο πεδίο με αυτό το οποίο είχαμε και στην αρχική τροπολογία της συμβαστική. Λοιπόν, η συμβαστική τροπολογία διαπιστώνει πως έχουν οι διάφορες δικαιοδοσίες και μας λέει ότι η δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, η δημιουργία δηλαδή ενός μηχανισμού ISDS, θα μπορούσε να λειτουργήσει ενάντια σε κάποιες εθνικές δικαιοδοσίες και προτείνει λοιπόν το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί με έναν νέο τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε επαγγελματίε δικαστές για τον νέο αυτό μηχανισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αναγκαστικά ένα μηχανισμό ISDS ο οποίος θα εντάσσεται σε αυτή τη συμφωνία. Επομένως, εμείς προτείνουμε όχι να αντιταχθούμε σε έναν μόνιμο νέο μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους. Αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής, το οποίο άλλωστε είναι και απόλυτα συμβατό με τη δεύτερη εκδοχή της συμβαστικής τροπολογίας 2 που μόλις εγκρίναμε προτείνουμε να μην συμπεριληφθεί μια συμφωνία επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους στα πλαίσια του TTIP, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα δικαστικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι η δεύτερη αυτή τροπολογία, η τροπολογία 16, έρχεται να διευκρινίσει περισσότερο την αρχική τροπολογία. Κύριε έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, να υποστηρίξω απλώ τα, αυτά τα οποία είπε η κυρία Περβόν Μπέχα. Ήταν απόλυτα σαφή. Για μας τα πράγματα είναι απόλυτα σαφή. Μιλάμε για μια διαφορετική πρόταση, η οποία όμως είναι απόλυτα συμβατή με την συμβαστική τροπολογία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 16. Στεμπάν. Ε, ε, Κύριος ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, οι προτινόμενες τώρα από τους συναδέλφους τροπολογίες έχουν να κάνουν με τις εθνικές δικαιοδοσίες, με τα εθνικά δικαστικά συστήματα. Ενώ εμείς αυτή τη στιγμή εγκρίναμε μια συμβαστική τροπολογία που αναφέρεται σε μια υπερεθνική δικαιοδοσία. Αυτή τη στιγμή εγκρίναμε μια συμβαστική τροπολογία η οποία δεν αποσαφηνίζει τα πράγματα. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή στη συμβαστική τροπολογία ποιε επιμέρου τροπολογίε καλύπτονται και ποιε όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από νομική πλευρά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ασαφή. Ψηφίσαμε μια συμβαστική τροπολογία και δεν ξέρουμε τώρα τι καλύπτει αυτή η συμβαστική τροπολογία. Εξ αρχή θα πρέπει τα πράγματα να αποσαφηνίζονται και όχι εκ των υστέρων να προσπαθούμε να δούμε τελικά τι καλύπτει η συμβαστική τροπολογία που μόλι συγκρίναμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η ερμηνεία των ομάδων, της ομάδας των σοσιαλιστών είναι αυτή που έδωσε η κυρία Μπερέζ. Υπάρχει νομική συμβατότης μεταξύ των δύο προτάσεων. Για τους ίδιους λόγους που παρουσιάστηκαν υπερασπιζόμαστε την ψηφοφορία της ε, τροπολογίας 16. Πρέπει να ψηφιστεί η 16. Elmar Brock. Also wenn ich den Ο κ. Elmar Brock. Mm. Διαβάζοντας τη νέα πρόταση βλέπω ότι υπάρχουν σχόλια, επικρίσεις που αφορούν τη διαδικασία. Αναφέρεται στους δικαστές κλπ. Εδώ λοιπόν εκφράζουμε περιορισμένη υποστήριξη για τα προτινόμενα ενώ η θέση της κυρίας Μπέρες είναι ε, απόρριψη. Έχει καλυφθεί λοιπόν η 16 διότι είναι ασύμβατη με το αίτημα που έχει υποβληθεί. Οι σοσιαλιστές δεν θα έπρεπε να είχαν στηρίξει την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άνεμανς. Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτή τη δήλωση, θα μπορούσα να πω και περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Δεν θα υπερψηφίσω τη δεύτερη εκδοχή της συμβαστικής αν γνώριζα ότι θα ψηφίζαμε την τροπολογία 16. Προτείνω απλώς να ψηφίσουμε τη δεύτερη εκδοχή της συμβιβαστική. Ε, ευχαριστώ. Ο κ. Καστάλτο. Η κυρία Μπρέσο. Ε, Εγώ θα ήθελα να προτείνω σε εκείνους που υπέβαλαν τη 17, 18 και 22 να αποσύρουν τις τροπολογίες του και έτσι δεν έχουμε το πρόβλημα τη μη νομιμότητα, τη συμβαστική που ψηφίσαμε. Θα ήταν η καλύτερη λύση. Uh, Άλλωστε, ο κύριο Σέπφλιν, εμεί το ΕΛΚ θα ε, ανησυχούμε πολύ για αυτό που συμβαίνει. Ας διακόψουμε για ένα δεκάλεπτο να το κουβεντιάσουμε άτυπα και μετά βλέπουμε κατά πόσο το ΕΛΚ είναι έτοιμο να συνεχίσει, είναι πρόθυμο να συνεχίσει με την ψηφοφορία. Πρόεδρος, πριν κάνουμε τη διακοπή που σχεδίαζα και εγώ, θα ήθελα να ακούσω όλους, να ακούσουμε τις απόψεις. Ο κύριος Καστάλντο είναι πρώτος. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με την ερμηνεία της συναδέλφου Μπέρες. Και να πω και κάτι. Στο κείμενο που λάβαμε εμείς, στη δεύτερη συμβαστική την εναλλακτική, η 16 δεν αναφέρεται πουθενά. Σαν τροπολογία που καλύπτει, αναφέρεται 17, 18 και 22, εν μέρη 24, 25, 23, αλλά 16 δεν αναφέρεται καν. Και κατά την άποψή μου γι' αυτό θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε για την ψηφοφορία και ξεμπερδεύουμε. Και τελειώνει η ιστορία. Διαφορετικά θα φύγουμε από εδώ. Οι πρόεδρος. Εκείνοι θέλουν να φύγουν, να σφύγουν. Λυπάμαι. Μου ζητήθηκε να κάνουμε και μια διακοπή 10 λεπτών για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και σαν πρόεδρος αυτό θα κάνω. Τη διακοπή. Διότι κάποιοι συνάδελφοι χρειάζονται μια διακοπή από ό,τι καταλάβα. Είναι... Εγώ προτείνω τη διακοπή για να βρούμε άτυπη συμβαστική. Θα δούμε αν θα δουλέψει, ίσως να μην τα καταφέρουμε. Αν λειτουργήσει καλώς, διαφορετικά, αν δεν βγει άκρη, δεν θα ήθελε το ΕΛΚ να συνεχίσει. Τουλάχιστον τα μέλη μου αυτό μου δείχνουν. Πρόεδρος, θα κάνω ότι δεν άκουσα το, αυτό που είπατε στο τέλος για τη διακοπή και για την προσπάθεια αυτό να κάνουμε. Λυπάμαι, ε, ναι, υπάρχουν κάποιοι που χρειάζονται διακοπή. Και ο εσωτερικό κανονισμό δεν μου απαγορεύει τη διακοπή σα. Δίνω 10 λεπτά και όχι παραπάνω. Ο Έλμαρ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ ζητώ η Επιτροπή μας να κάνει εξακρίβωση, να επαληθεύσει, να δει μήπως Μία δεύτερη συμβιβαστική θα μπορούσε να υποβληθεί. Νομίζω ότι έγινε κάποιο είδος πραξικόπημα που έγινε. Πρωτοφανές. Είμαι εδώ χρόνια και ποτέ δεν είδα τέτοιο τρόπο διαδικασίας. Δεν είναι σωστός ο τρόπος αυτός. Πρόκειται περί πραξικοπήματος που εγώ δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ιδού λοιπόν. Γι' αυτό θα κάνουμε διακοπή 10 λεπτών για εκείνους που θέλουν να συνομιλήσουν. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν το κουβεντιάζουν. Θα τα πούμε ξανά σε 10 λεπτά. Ελπίζω να είχατε αρκετό χρόνο για να συζητήσετε. Ας ξεκινήσουμε με τον εισηγητή. Ποια είναι η άποψή του για την τροπολογία 16. Δεν αναφέρεται και έτσι στη συμβαστική και μπορούμε να ψηφίσουμε, να την ψηφίσουμε. Αυτό προτείνω να κάνουμε σαν εισηγητής. Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη εδώ δεν συνάδει με την καλή συμπεριφορά. Εγώ είδα τη συμβαστική σήμερα το πρωί σαν εισηγητής. Ελπίζω ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό και δεν θα ξαναγίνει αυτό που συνέβη σήμερα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όταν έλαβε την τροπολογία η γραμματεία, τη συμβαστική τροπολογία, η πληροφορίε ήταν ότι και ο εισηγητή έλαβε τη συμβαστική. Δεν μπορεί να κατηγορεί τη γραμματεία γι' αυτό. Το δεύτερο. Κάτι έγινε στο σύστημα που δεν λειτουργήσε σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να σας πω. Διαβάζω, ξαναδιαβάζω και η τροπολογία ξεκινά. Λέει, στόχος να αντιταχθούμε στην εισαγωγή του μηχανισμού ISDS στο TTIP. Αυτό δεν είναι αντίθετο με τη συμβαστική. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι αντίθετη η συμβαστική που ψηφίσαμε. αναφέρεται σε μεγαλύτερη φιλοδοξία να έχουμε μια μόνιμη λύση. Το πνεύμα είναι εντελώ διαφορετικό. Στη συμβαστική επιδιώκουμε μόνιμη λύση. Κάτι δύσκολο. Στο τέλος του δρόμου. Εδώ έχουμε τη συμβαστική που ξεκινά με κάθετη αντίθεση συμπεριλήψη του ISDS στο TTIP. Αν αυτό είναι κάτι συμβατό, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου εκφράστηκαν και άλλες απόψεις. Και είχατε δικαίωμα να ζητήσετε ψήφο παρά τα όσα σας είπα. Έχουμε και τη δήλωση του εισηγητή που εξετάζει με ειλικρίνεια τον δεχόμενο να υπάρχει κάτι που δεν καλύπτεται από τη συμβαστική που ψηφίσαμε. Εγώ δεν συμφωνώ όμως και λυπάμαι που το λέω έχουμε την εξής επιλογή. Μπορούμε να ψηφίσουμε αν θεωρούμε ότι είναι συμβατή ή όχι. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση όσον αφορά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας. Γι' αυτό. Εγώ είμαι κατά. Εσείς είστε κατά της προσέγγισης. Είσαστε αντίθετοι με την ε, ISDS που είναι η θέση της ΑΦΚΟ. Εγώ είπα ότι δεν είναι ασύμβατη και ο εισηγητής. Κατά την άποψή μας να ψηφίσουμε. Αν προτιμάτε εσείς να ζητήσετε εκ των προτένων θέλετε να ψηφίσουμε ή όχι, έχετε δικαίωμα. Ναι, θα το κάνω, λέει η Πρόεδρος. Ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά θα το θέσω. Η Περβάμς Περές θα ψηφίσει. Θα δούμε αν είναι παραπάνω, θα δούμε στην οθόνη αν είναι κάποιος παραπάνω στην ψηφοφορία. Δεν έχετε κάρτα εσείς. Πώς ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε πολλούς. Πρέπει να μετρήσουμε τους σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές, σηκώστε τα χεράκια, συγγνώμη, τα χέρια σας για να δούμε πώς είσαστε. Έξι. Είναι το όριο, εντάξει. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την περβάνηση Ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε, να το προσθέσουμε Ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε την τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε την 16. Μετάει κάποιος. Είναι σαφής η πλειοψηφία πιστεύω. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Κατά τις ψηφοφορίες, Κατά τις ψηφοφορίες της 16 ποιος είναι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 16. όλες οι άλλες που θεωρούνται ως καλυμμένες από την συμβαστική δεν θα ψηφιστούν και πρέπει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Κάποιος ζήτησε ονομαστική. Ψηφίζουμε την 16 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Χωρίς την Περβάνς έχουμε ήδη 25. Με την Περβάνς είμαστε 26 και έχουμε μόνο 25 μέλη. Α, εντάξει. Okay, okay. Okay. So, so it's 14 to... 14 υπέρ 11 κατά. Ευχαριστώ. 14 to 11. 14 to 11. Τροπολογία 28. Υπέρ της 28. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ Κατά. Έλεγχος για την 30. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Figures. Colleagues don't see the figures.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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32, τελευταίο τμήμα της τροπολογίας είναι συμβατό με συμβαστική 3. Ψηφίζουμε το τελευταίο τμήμα που ξεκινά και ζητά μέχρι δημόσιο. Ποιος είναι υπέρ αυτού του τμήματος της τροπολογίας. Κατά. Αποχές απορρίπτεται νομίζω. Έλεγχος για 32. Άρχεται η ψηφοφορία, ο έλεγχος για την 32. Απορρίπτεται μεγάλη διαφορά. 17 κατά, 7 υπέρ. Μεγάλη διαφορά. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται θάρρο. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά έλεγχος για την 52 Έχουμε ένα μέλος, ένα μέλος του ΕΡΚ παραπάνω. Θέλουμε ένα μέλος του ΕΛΚ λιγότερο. Τώρα όλα είναι εντάξει. Μην κινηθείτε καν. Μην αναπνέτε. Πέρας φοφορία. απορρίπτεται. 53 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία υπάρχει αίτημα για νομαστική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο Καλώς τώρα, είμαστε σωστοί τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, 2 εποχές. Τελειώσαμε, θα τα ξαναπούμε στις 3. Ευχαριστούμε πολύ, καλή όρεξη.